Mesdames et messieurs, bonjour Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην συνάντηση αυτή όπου θα ακούσουμε τα συμπεράσματα από τα εργαστήρια της αγοράς. Ελπίζω ότι θα είναι καρποφόρο το πρωινό, συγκεκριμένο και θα μας ε, δώσει τροφή για να δουλέψουμε στη συνέχεια εδώ εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα το πρωί θα ακούσουμε τα συμπεράσματα των τριών εργαστηρίων και θα ακούσουμε και τα συμπεράσματα της διάσκεψης της συνένεσης. Εδώ οι 20 πολίτες που συμμετείχαν ε, σε αυτό το εργαστήριο θα μας παρουσιάσουν τα συμπεράσματα των ε, εργασιών τους τις δύο Μέρε που μα πέρασαν, γιατί αυτοί δούλεψαν λίγο παραπάνω από του άλλου. Στι 11 θα κάνουμε διάλειμμα για καφέ. Ο κύριο Ρούτσεκ και εγώ θα μπορέσουμε έτσι να πάμε να παρουσιάσουμε στον τύπο, στα μέσα ενημέρωση, τον καρπό των εργασιών σα. Και μετά θα επανέλθουμε για να εμβαθύνουμε περισσότερο στη συζήτηση, για να προσθέσετε, εφόσον θέλετε, ό,τι νομίζετε στα συμπεράσματα και στη συνέχεια να κλείσουμε έτσι τη συνάντηση αυτή της αγοράς. Και τότε η χοροδία υπό το φως του φεγγαριού ο Κλέρ Δελαλούνε θα μας ε, παρουσιάσει και λίγο μουσική με κάποιο τραγούδι. Έχετε μπροστά σας τα έγγραφα στα γαλλικά με τα συμπεράσματα. Τα αγγλικά θα έρθουν όπου να είναι. Μέσα στο επόμενο μισάωρο θα έρθουν. Τυπώνονται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ εξάλλου και τους μεταφραστές και όλους όσοι δούλεψαν χτες αργά το βράδυ και σήμερα το πρωί για να μεταφράσουν τα έγγραφα αυτά. Α, δεν τα έχετε μπροστά σας. Ε, θα έρθουν όπου να είναι. Μην φοβάστε, όπου να είναι θα τα έχετε μπροστά σας. Νόμιζα ότι είχαν ήδη μοιραστεί. Όπως και να έχει το πράγμα. Πάντως, προφορικά θα τα διαβάσουμε, οπότε μέσω της διερμηνίας θα τα ακούσετε στη γλώσσα σας. Οπότε έτσι θα τα καταλάβετε. Ξεκινάω λοιπόν από την πρώτη ομάδα εργασίας που είχε ως θέμα την οικονομική και δημοσιονομική κρίση και νέα φτώχεια. Πρόεδρος είναι η κυρία Τζιν Λάμπερς, ευρωβουλευτής. Η κυρία Χίλντα Φιγερέρο και ο κύριος Σπινά, επίσης ευρωβουλευτές, ήταν συνεισηγητές. Η κυρία Φιγκερέρο θα πάρει τώρα το λόγο. Πρέπει να πάρει το αεροπλάνο σε λίγο και θα χρειαστεί να φύγει, οπότε θα ξεκινήσω με εκείνη. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε λοιπόν εδώ σήμερα το πρωί και θα συμπληρώσει ο διπλανός σας, έτσι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Στην ομάδα εργασίας μας είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Συζητήσαμε για την φτώχεια, για τις αιτίες της φτώχειας, για την κρίση. Μιλήσαμε επίσης και για τα μέτρα που ε, προτείνουν οι διάφορες οργανώσεις για να αντιμετωπιστεί ακριβώς αυτή η κατάσταση. Ακούσαμε και διαμαρτυρίες για την αύξηση της φτώχειας και για το ότι δεν υπάρχουν αρκετά μέτρα ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Mm. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρίως, θα επιληθούμε του μηνύματος αυτού. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε κάποια μέτρα. Πρέπει να καταλάβουμε σε τι κατάσταση ακριβώς ζούμε εμείς σήμερα. Και πρέπει να προσπαθήσουμε πάση θυσία να βρούμε κάποιες λύσεις. Πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που ζουν μέσα σε αυτή την κατάσταση. Εξού και η πρότασή μας να δημιουργηθούν κάποιες ομάδες εργασίας. Ο συνάδελφος, συνεισηγητής, πιο συγκεκριμένα θα σας μιλήσει για τις προτάσεις μας. Κάποιες οργανώσεις που ασχολούνται με τα κοινωνικά θέματα υπέβαλαν προτάσεις και θα σας τις παρουσιάσουμε σε λίγο. Ζήτησαν βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσουν, να επιμείνουν ώστε να δοθεί κάποια συνέχεια στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου μας για παράδειγμα. Βέβαια δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα, δεν δώσαμε απαντήσεις σε όλα. Σίγουρα όμως το Κοινοβούλιο και οι Ευρωβουλευτές πρέπει να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα το τι συμβαίνει. Χρειάζεται ένα ελάχιστο κειμένο εισόδημα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια νομοθετική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαία κατά τη γνώμη μας. Χρειαζόμαστε μια πρόταση. Δεν έχουμε ακόμα νομοθετικές προτάσεις. Εγώ προσπαθώ να δουλέψω πάνω σε αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε μια τέτοια θέση. Όμως δεν ανελήφθη καμία πρωτοβουλία. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορεί να υποβάλει μια τέτοια πρωτοβουλία κανένα άλλος. Πάντως, οικονομική και κοινωνική συνοχή, ευημερία των πολιτών, αξιοπρέπεια των ανθρώπων, αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Και πρέπει οι πολιτικοί να λαμβάνουν υπόψη τους ανθρώπους και πρώτα να βλέπουν τι αντίκτυπο θα έχει η πολιτική που προτείνουν και μετά να την ε, κάνουν πράξη. Θέλουμε οικονομικά μέτρα και αποσύνδεση, μάλλον και να μην υπάρχει αποσύνδεση της οικονομικής πτυχής από τη μία και της κοινωνικής από την άλλη. Όχι, αυτά τα δύο πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Επικρίναμε πάντω την κατάσταση στην ομάδα εργασίας μας ξανά και ξανά. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ξέρουμε πάντα ένα οικονομικό μέτρο τι κοινωνικές συνέπειες θα έχει με την αύξηση της ένδειας, της ανεργίας, ε, των κακοπληρωμένων επαγγελματικών θέσεων δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Έχουμε μια κατάσταση ένδειας, φτώχειας που επιδεινώνεται συνεχώς και έχουμε και νέες μορφές μάλιστα φτώχειας. Έχουμε τους φτωχούς εργαζόμενους. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού, τους νέους, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα θέματα αυτά θα τα συζητήσουμε τους επόμενους μήνες στα πλαίσια της κοινωνικής ασφάλισης. Γι' αυτό και πιστήσαμε την προσοχή σε μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις ώστε και ηλικιωμένοι να ζουν με αξιοπρέπεια. Έπειτα υπάρχει το θέμα της πρόσβασης στις κοινοφελείς υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες, και γενικού ενδιαφέροντος. Ο συνάδελφος συζητητής θα σας τα πει όλα αυτά με λεπτομέρειες. Θα σας παρουσιάσει και τις προτάσεις που υπέβαλαν οι διάφορες οργανώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ελπίζω επιτέλους να έχετε καταλάβει ότι αυτή η δυσαρέσκεια, αυτή η απογοήτευση πρέπει να διοχετευτεί, πρέπει να φτάσει στις κυβερνήσεις που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ώστε να ληφθούν οικονομικά και κοινωνικά ε, μέτρα, καλύτερα από αυτά που έχουμε μέχρι τώρα. Εγώ προσωπικά αυτή την έκκληση κάνω, αυτή την απογοήτευση διοχετεύστε την, καταδικάστε αυτά που συμβαίνουν. Αυτό είναι το μήνυμά μου από την απογοήτευση που ζει ο κόσμος διαπιστώνοντας την επιδείνωση της ένδυας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο άλλος συνεισηγητής και είδατε ότι σε κάθε εργαστήρι υπάρχει ένας εισηγητής από την Ευρωβουλή και ένας από τα συνδικάτα ή από τις οργανώσεις κτλ. Έχετε το λόγο κύριε. Από ό,τι μου είπαν μπορώ να μιλήσω και Ολλανδικά, έτσι. Και αυτό θα κάνω, θα μιλήσω Ολλανδικά. Έχω εδώ τη γραπτή έκθεση της ε, ομάδας μας. Το είδα ε, σήμερα το πρωί. Σίγουρα είναι δύσκολο να σας τα πω όλα, αλλά έτσι απ' έξω θα προσπαθήσω να σας και γραφήσω τα κυριότερα σημεία. Πρώτα απ' όλα. Για το θυμό που νιώθει ο κόσμο εξαιτία τη κοινωνική κατάσταση που ζει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να βρει έναν τρόπο να βοηθήσει ώστε ο θυμό αυτό να διοχετευτεί, να γίνει ορατό, να προβληθεί και να υπάρξει μια μεγάλη συζήτηση για τι αιτίε που οδηγούν σε αυτήν την δυσάρεστη κοινωνική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Να εντοπιστούν οι αιτίε αν θέλουμε να βρούμε και λύσεις. Ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο κατάλληλος χώρος για να οργανωθεί μια τέτοια συζήτηση, ώστε να έχουμε νέες ιδέες, νέα παραδείγματα συνύπαρξής μας ε, στις κοινωνίες μας. Δυστυχώς οι λύσεις που έχουμε μέχρι τώρα δεν είναι ικανοποιητικές. Στην ομάδα εργασίας επίσης ζητήσαμε ε, περισσότερη κοινωνική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ξεκάθαρο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει την πρωτοβουλία για να κάνει τέτοιε, δεν έχει δικαίωμα πρωτοβουλία για τέτοιε προτάσει η Επιτροπή. Αλλά εμεί μπορούμε να πιέσουμε για να αναλυθούν τέτοιε πρωτοβουλίε από την Επιτροπή. Νομοθεσία λοιπόν θέλουμε επίση στον τομέα του χρέου. Και προκειμένου να προλάβουμε ε, υπερβολικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η χρέωση των πιο ευάλωτων πληθυσμών. Όπως είπε και η κυρία Φεγγερέρο, η νομοθεσία πρέπει να υπάρξει και σε άλλους τομείς για να προστατευτούν τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα. Πολλές φορές δεν είναι γνωστό στον κόσμο ότι το Κοινοβούλιο σήμερα έχει περισσότερες εξουσίες από ό,τι είχε κατά το παρελθόν και για το ευρώ και για τις κοινωνικές επιπτώσεις. Γι' αυτό και λέμε ότι μπορούμε να πιέσουμε για νομοθεσία. Έπειτα, πολλοί συμμετέχοντες μίλησαν για την μέθοδο ανοιχτού συντονισμού. Είπαν ότι η μέθοδος αυτή πρέπει να ενισχυθεί στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στην καταπολέμηση της ε, ένδυας και να φροντίσει για αντίστοιχη πολιτική εδώ. Ζητήθηκε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να θέσει πιο ξεκάθαρα τα δικά του θέματα όσον αφορά την ένδυα προς τα άλλα κοινωτικά όργανα. Ότι θα πρέπει δηλαδή τα άλλα ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα να μας ακούνε περισσότερο, να μας λαμβάνουν υπόψη τους, να λαμβάνουν υπόψη τους τι ζητάει το Κοινοβούλιο και να δίνουν συνέχεια σε αυτό. Υπάρχει ένα θέμα που εγώ γνωρίζω καλά και για το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα έκανε μια γραπτή δήλωση με την οποία ζητάει το Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να φροντίσουν να δημιουργηθεί μια ομάδα για να εξετάσει όλα αυτά τα ζητήματα το θέμα της ένδυας, τη, του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος κλπ. κλπ. Έπειτα μιλήσαμε και για τον λεγόμενο τέταρτο κόσμο, για τους φτωχούς δηλαδή στις πλούσιες χώρες. Είναι και αυτό ένα θέμα που έχει μεγάλη σημασία για μας. Θέλουμε να ακούσουμε τους ανθρώπους που έχουν εμπειρία όμως σε αυτά τα ζητήματα για τη φτώχεια. Γι' αυτό και σας φωνάξαμε εδώ, που ζουν στη φτώχεια. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια καλύτερη πολιτική. Δεν είναι κάτι απλό βέβαια στην πράξη, το ξέρουμε. Στη συνέχεια. Υπήρξαν και άλλα θέματα. Το θέμα του προϋπολογισμού. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να φροντίσουμε να καλύψουμε τα κενά που έχουμε σχετικά με την ένδια. Δεν γνωρίζουμε μερικές φορές καλά το πρόβλημα και δεν μπορούμε να φροντίσουμε να, αντικατα... να αντικατοπτριστεί και στον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να βοηθήσουμε τον κόσμο που ζει στη φτώχεια. Συζητήσαμε για την μετανάστευση επίσης ε, από την Ανατολική Ευρώπη προς τη Δυτική Ευρώπη. Εκτός αυτού ακούσαμε και άλλα πράγματα σημαντικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν να κάνουν με την πολιτική μας. Ότι η φτώχεια είναι πολυδιάστατη, ότι πρέπει να τη δούμε από διάφορες πλευρές, ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το οικονομικό από το κοινωνικό σκέλος, ότι είναι πολλοί οι φορείς που πρέπει να συμμετέχουν στη λύση και ότι ίσως θα πρέπει να υπάρχουν ομάδες στόχοι με τους οποίους να ασχοληθούμε ιδιαίτερα, πιο ευάλωτοι δηλαδή παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι. Και κάτι άλλο που χτες ακούσαμε είναι ότι πρέπει να χτίσουμε πάνω στα κεκτημένα μας. Γιατί δεν είναι ότι δεν υπάρχει και τίποτα. Δεν είναι ότι δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα μέχρι τώρα. Υπάρχουν κάποια πράγματα. Πάνω σε αυτά πρέπει να φροντίσουμε να χτίσουμε για να πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Και άλλα πράγματα στη γραπτή έκθεση αναφέρονται. Τώρα εγώ δεν σα τη διάβασα. Νομίζω ότι σας έκανα μια πολύ καλή περίληψη. Σας είπα ποια ήταν τα πιο σοβαρά, τα πιο συγκεκριμένα και σημαντικά θέματα που συζητήσαμε και στα οποία καταλήξαμε χτες. Σας ευχαριστούμε κύριε σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Όντως η έκθεση υπάρχει και μοιράζεται αυτή τη στιγμή αλλά εξίσου σημαντικό είναι να δούμε και με τι ύφο έγινε η συζήτηση ε, στην ομάδα. Η, η, η οργή αυτή, η δυσφορία, η κοινωνική θα έπρεπε πολύ σωστά να περάσει ως πνεύμα στο Ευρωκοινοβούλιο μας. Θα έχουμε τη συζήτηση μετά. Αν όμως κάποιος μέλος από το ε, συνεδρίαση αυτή από το ατελείο, όπως το λέμε αυτό, θέλει αυτή τη στιγμή να προσθέσει κάτι καλός, Αλλιώ θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Έτσι κι αλλιώ όμω μετά τη διακοπή του διάλειμμα για τον καφέ θα, θα επανέλθουμε για συζήτηση. Το νούμερο 342 μου ζήτησε το λόγο. Κυρία μου, έχετε το λόγο. Σερ Τζόνσον από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Φτώχειας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σύνοψη. Ήταν ένα σεμινάριο το οποίο κάλυψε καλά το θέμα, ιδιαίτερα για την αγανάκτηση και την οργή για αυτά που συμβαίνουν και την ανάγκη για δράση. Και υπάρχουν μερικά σημεία που ίσως δεν λήφθησαν υπόψη συγκεκριμένα. Κάναμε μερικά, μερικά συγκεκριμένα αιτήματα σχετικά με το τι θα μπορούσε να κάνει το Ευρωκοινοβούλιο. Π.χ. οι αιτίε της κρίσης, η κοινωνική επίπτωση της κρίσης, το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Ξεκινώντας μια συζήτηση, έχω μια αξιολόγηση επιπτώσεων που την έκανε η Κομισιόν, από ό,τι ξέρουμε το Κοινοβούλιο δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή. Δεύτερον, η Ευρώπη 2020. Αυτό που συμβαίνει τώρα γίνεται φυσικά μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης 2020. Έχουμε μια νέα έκθεση πρόοδου, την διάφορες πλατφόρμες ευελιξίας, στόχους κατά της στόχιας. Θέλουμε το Κοινοβούλιο να το δει ως συνολικό πακέτο, γιατί για μας η οικονομία υπονομεύει τα κοινωνικά. Έχουμε μια έκθεση που λέει ότι ε, φορολογική ε, εξυγίανση, μείωση όσο πιο γρήγορα γίνεται των των δημοσίων ελλημάτων, ποιο είναι ο ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου. Κατά τη γνώμη μα, θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα εργασία στο Ευρωκοινοβούλιο που να παρακολουθεί συνολικά το θέμα Ευρώπη 2020 και όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να παίρνουν μέρο. Μετά πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση με εθνικά επίπεδα, να υπάρχουν εθνικέ πλατφόρμε κατά τι φτώχεια, εθνικέ στρατηγικέ κατά τη ε, ε φτώχεια, ε, του μη κοινωνικού αποκλεισμού για αυτούς που ζουν τη φτώχεια και μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Δύο προτάσεις. Πρώτον, επίπεδο ένωσης. Δεύτερον, εθνικό επίπεδο για να βγουν επιτέλους κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα από την αγορά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για τις προτάσεις αυτές. Τι σημειώνω, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μετά, τι συνέχεια να δώσουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Άλλα σχόλια από αυτούς που πήραν μέρος σε αυτό το πρώτο ατελείο, όπως το λέμε. Ο κύριος στο νούμερο 65 από την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή. Είμαι μέλος της Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής από τη Ρουμανία. Εκπροσωπώ μια συνδικαλιστική οργάνωση. Θα συνεχίσω στα ρουμανικά. Ευχαριστώ. Πολλά ενδιαφέροντα πράγματα ακούστηκαν νομίζω και στις τρεις ομάδες εργασίας. Είναι ξεκάθαρο ότι οι κυβερνήσεις των χωρών μελών πρέπει να παρεμβαίνουν με μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας. Ναι, αυτό όμως από την άλλη δεν πρέπει να σημαίνει ότι αφήνουμε στην πάντα κάτι άλλο πολύ σημαντικό που είναι το εξής. Τα προβλήματα του οικονομικού συστήματος, του νεοφιλελεύθερου συστήματος, ενός συστήματος που επικρατεί στις περισσότερες χώρες μέλη, είναι και αυτό κάτι που πρέπει να δούμε και που πρέπει να αλλάξει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί το είδος αυτό της κρίσης που μας έχει οδηγήσει σε τόσα προβλήματα και που αυξάνει τον αριθμό των ανθρώπων που υποφέρουν από φτώχεια δεν πρέπει να επαναληφθεί. Εγώ συμμετέχω όντως στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και πρέπει να σας πω ότι χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα όργανα που δημιουργούνται για παράδειγμα, οι αρχές για την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος ή για την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, η αρχή για τις δημοσιονομικές αγορές. Όλα αυτά τα όργανα πρέπει να έχουν πραγματική εξουσία ελέγχου και εποπτείας εκεί όπου είναι αρμόδια. Όπως πολύ σωστά έλεγε και ο, ο Λούτσεκ, Ορισμένοι, ορισμένες χώρες μέλη αντιτίθεται. Δεν τον θέλουν αυτό τον έλεγχο, αυτή την εποπτεία. Όμως, αν δεν διορθωθούν τα προβλήματα που οφείλονται στον οικονομικό μηχανισμό, τότε η καταπολέμηση της φτώχειας δεν θα οδηγήσει πουθενά. Δεν θα πετύχει. Και όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν θα πετύχουν. Ενώ αντίθετα πρέπει να στηριχτούν Αυτά τα όργανα λοιπόν που δημιουργούνται πρέπει να είναι όργανα που έχουν πραγματική εξουσία ελέγχου και πραγματική δύναμη για να καταπολεμήσουν τι αρνητικέ επιπτώσει του οικονομικού συστήματο. Τέτοιε κρίσει, σαν και αυτή που έχουμε σήμερα, δεν πρέπει να επαναληφθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακόμη μία παρέμβαση και μετά θα προχωρήσουμε στο δεύτερο εργαστήρι. Εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σε όλους. Ισπανικά θα μιλήσω, λέει ο Για την ομάδα εργασίας ε, αριθμός 1. Ακούσαμε από τον εισηγητή ότι πρέπει να γίνει δουλειά στις χώρες μέλη, ότι δεν φτάνει εδώ να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας και στις χώρες μας. Και εμείς είπαμε ότι δουλεύουμε στις χώρες μας και ότι η αγανάκτηση έρχεται από τις χώρες μας ακριβώς και φτάνει σιγά σιγά εδώ. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν διαμαρτυρόμαστε, ότι δεν αγωνιζόμαστε, δεν ε, δείχνουμε την οργή και την αγανάκτησή μας στις χώρες μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφόσον ασχοληθεί και αυτό με αυτά τα θέματα, αυτό μας βοηθάει σε αυτά που κάνουμε εμείς στις χώρες μας, με τις κυβερνήσεις μας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συζητήσει τις επιπτώσεις, τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, όχι μόνο τις οικονομικές, με νούμερα για τους δημοσιονομικούς οργανισμούς, για το πώς επηρέασε αυτό και το βιομηχανή κτλ. Δεν λέω και αυτό είναι σημαντικό και αναγκαίο, αλλά πρέπει να συζητήσει και το πώς επηρεάζονται οι άνθρωποι. Διότι οι ευρωπαϊκέ χώρε είναι σημαντικέ, αλλά και οι ευρωπαίοι πολίτε είναι σημαντικοί. Γι' αυτό να δούμε η κρίση αυτή πώ επηρεάζει τον πολίτη. Τι συμβαίνει με αυτόν, τι έχει γίνει με του ε, ανθρώπου στην κάθε χώρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν ζητάμε να μελετήσει την κοινωνική επίπτωση που έχει η κρίση, να παρακολουθήσει επίση με τη στρατηγική 2020 που θα μα οδηγήσει. Συμφωνώ με αυτά που είπαν εκεί προλαλήσαντες εδώ. Είναι αναγκαίο. Γιατί η συζήτηση αυτών των πραγμάτων εδώ μας βοηθάει εμάς στη δουλειά που κάνουμε στις χώρες μας, στην κοινωνία των πολιτών. Δουλεύουμε εκεί και αγωνιζόμαστε εκεί, ώστε οι επιπτώσεις της κρίσης να είναι όσο γίνεται λιγότερο σοβαρές για τον πολίτη. Euh, Ακόμη μια σύντομη παρέμβαση. Θα είμαι σύντομος. Χθες, λέγομαι Φιλίπ Ρόγε, είχα προτείνει στην ομάδα εργασία μου η Ευρωβουλή να νομοθετήσει για ένα νομικό πλαίσιο για τις ε, πιστοτικές οργανώσεις, για τα πιστοτικούς οργανισμούς που προσφέρουν δάνεια στην κατανάλωση. Δεν περιλήφθηκε αυτό ε, στην σύνοψη του εισηγητή. Επίσης για την μετεκατάσταση των επιχειρήσεων προσφέρουν απασχόληση. Εκεί δηλαδή που πηγαίνουν σε χώρες που έχουν χαμηλές κοινωνικές εισφορές. Και έτσι προκαλείται απώλεια κυρίως ε, θέσεων στην οικοδομή. Και επομένως αυτό προκαλεί πάλι με τη σειρά του φτώχεια. Σας ευχαριστώ. Τώρα έρχεται το εργαστήρι παριθμό 2 που είχε για θέμα κρίσεις και μεταναστευτικές ροές με επικεφαλής τον κύριο Νταρντέν και δύο συνεισηγητές Βαρντού και Βενχάγεν η κυρία Μπέναραμπ πρώτη Ευχαριστώ πρώτα όλες και όλους που συμμετέσχουν θα δώσω αμέσω τον λόγο αν επιτρέπετε στον συνεισηγητή μου μέσα στα πλαίσια των οδηγιών που είχαμε και των αρμοδιοτήτων της Ευρωβουλής συντάξαμε τις εξής προτάσεις. Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών απευθύνουν έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών σε σχέση με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αβέβαιες θέσεις για να επανέλθει στις αξίες πάνω στις οποίες ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέσα στα πλαίσια των αρμοδιότητων που προσφέρει στην Ευρωβουλή ε, η συνθήκη της Λισαβόνα, να σεβαστεί τις διατάξεις της συνθήκης της Γενέβης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του θεμελιώδη χάρτη, του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων δηλαδή, καθώ και των άλλων ε, διεθνών συνθήκων και διατάξεων που επιβάλλονται. Να δεστεί μια βάση η οποία θα εγγυάται την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των μεταναστών χωρί άνηση μεταχείριση, χωρίς διάκριση οικονομική, κοινωνική και να ξαναρχίσει η συζήτηση για το δικαίωμα ασύλου προκειμένου να οριστεί με ανθρωπιστικό τρόπο. Να υπάρξει ένα οικονομικό πλαίσιο 2014-2020 με βάση τη στρατηγική της 2020 και τους στόχους χιλιετίας για την ανάπτυξη. Να δούμε πώς είναι δυνατόν να υπάρξει καλύτερη συμπληρωματικότητα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης. Έτσι ώστε οι προτεραιότητες Ένωσης για θέματα μετανάστευσης να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες πολιτικές και προϋπολογισμούς. Καλούμε επίσης το Ευρωκοινοβούλιο να ζητήσει από την Κομισιόν να ξεκινήσει μία συζήτηση με όλα τα κράτη-μέλη και την κοινωνία των πολιτών για την πρόθεση της αμοιβέ και συνθήκες εργασίας αξιοπρεπής. Να ενθαρρυνθεί η δημιουργία δικτύου για την κοινωνία των πολιτών σε θέματα ενσωμάτωσης του μετανάστη, έτσι ώστε να ευνοηθεί η συμμετοχή των εκπροσώπων του σε αυτές τις δραστηριότητες και πιο συγκεκριμένα μέσω ακροάσεων και συζητήσεων και να χρησιμοποιηθεί η εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει με βάση τις ε, πολιτικές για τη μετανάστευση στην Ένωση. Έβδομο, να ευνοηθεί η αναγνώριση των πανεπιστημιακών ε, διπλωμάτων και επαγγελματικών προσόντων πολιτών τρίτων χωρών έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας της Ένωσης. Αυτή η αναγνώριση να τυποποιηθεί με υπογραφή συμφωνιών με τις τρίτες χώρες. Να διασφαλιστεί καλή συνεργασία μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και των εθνικών βουλευτών με βάση το πρωτόκολλο για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ένωση που είναι παράτημα της συνθήκης και τη λειτουργία της Ένωσης. Κατά πολέμη συνέχιση της μάχης κατά πάσης μορφής ρατσισμού και άνηση μεταχείριση στην Ευρώπη για την πρόθεση της ενσωμάτωσης των μεταναστών με, ε, με μια ορολογία που θα είναι ευνοϊκή στον γίνον αποδεκτή από τα μέσα ενημέρωση και την κοινή γνώμη οι μετανάστες και γενικά για τις πολιτικές κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών. με πρόθεση μια ανοιχτή έννοια, τη ιδιότητας του πολίτη που να καλύπτει όλους τους πολίτες, τους νόμους και τους μη νόμου. Να φροντίσουν για την εφαρμογή ενός πλαισίου κατάγγελο για την εθελοντική δράση στην Ένωση, έτσι ώστε ο εθελοντισμός να βοηθήσει την προσπάθεια συμμετοχής στις Κοινωνικέ ενέργειε. Τέλο να ενθαρρυνθεί το Ευρωκοινοβούλιο να υπογράψει τη γραπτή δήλωση 086 των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά του μετανάστε εργαζόμενου. Και τέλος, καλούνται τα κράτη-μέλη να φροντίσουν για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της, ε, του Ευρωπαϊκού Χάρτη των ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε ότι ε, καλύψαμε σωστά ε, ε, τα πορίσματα της ομάδας εργασίας μας στο εργαστήριο. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ τους δύο συνηγητές για τις πολύ συγκεκριμένες αυτές συστάσεις και πραγματικά έρθήκατε στο ύψος των όσων συζητήθηκαν στο εργαστήρι σας. Άλλος κανείς επιθυμεί να παρέμβει, εσείς κυρία μου στο 350. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές γιατί πραγματικά εξήγησαν ακριβώς τα όσα συζητήσαμε. Μια ανησυχία που έχω, δεν ξέρω ίσως να εμφανίζεται κάπου αλλού μέσα στις συστάσεις, σχετικά δηλαδή με το δικαίωμα των προσώπων που ζητούν άσυλο. Δεν ξέρω αν είναι μέσα, είναι το, το, το ζήτημα του σωματεμπορίου. Το λέω αυτό για να είναι σίγουρο ότι κάπου, κάπου έχει περιληφθεί. Αυτό το πρόβλημα δηλαδή. Η κυρία Μπεναράμπ. Ναι, δεν το έχουμε βάλει, αλλά έχετε δίκιο, θα το περιλάβουμε, θα το, θα το προσθέσουμε. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Η... Ο κύριος Τζουλιάνο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ είμαι μέλο τη Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή και είχα την τιμή να συμμετέχω στην ομάδα αυτή εργασία και μίλησα κιόλα. Πράγματι, καλύπτονται όλα τα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πάω πέρα από την αναγκαία σύνθεση, η οποία σωστά έγινε όλων αυτών των σημείων για να αναφέρω ένα τμήμα της συζήτησής μας που τη βρήκα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και αποκαλύπτεται στο σημείο 3 και στο σημείο 10 μια ανοιχτή έννοια της ιδιότητας του πολίτη. Πολύ σωστή έγινε η σύνθεση στο σημείο αυτό για την έννοια του μετανάστη εργαζόμενο. Γιατί υπάρχει ένας ορισμός αλλά είναι υπεραπλουστευμένος. Οι μετανάστες εργαζόμενοι είναι πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται προς την Ένωση, στον χώρο της Ένωσης για εργασία. Αντίθετα, η έννοια του μετανάστη εργαζόμενου πρέπει να καλύπτει και τις μεταναστευτικές ροές που συμβαίνουν μέσα στις χώρες Ένωσης, από χώρα σε χώρα της Ένωσης και στο εσωτερικό της κάθε χώρας. Γιατί οι μετανάστες εργαζόμενοι δεν είναι μόνο δεν θα πρέπει να αναφέρεται μόνο στην ελεύθερη κυκλοφορία του εργαζόμενου, θα πρέπει να αναφέρεται στην κοινωνική ταυτότητα, στο δικαίωμα του πολίτη. Επαναλαμβάνω, κοινωνική ταυτότητα που έχει σχέση με τη δυνατότητα κάποιου να βρει δουλειά. Πάμε χάρη οι πολλοί Ρουμάνοι που υπάρχουν στην Ιταλία για τους οποίους ακόμα παρόλε τις προσαρμογές της νομοθεσίας που έγιναν δεν υπάρχει κοινωνική προστασία προβλέπονται για τους ε, Ιταλούς πολίτες αλλά όχι για αυτούς που βρίσκονται εν μετακινήσει. Επαναλαμβάνω, αυτή η έννοια της μετανάστευσης πρέπει να συνδέεται στενά με την κοινωνική ταυτότητα και το δικαίωμα του πολίτη. Η έκθεση, το ξαναλέω, είναι άριστη. Ήθελα μόνο να επισημάνω κάτι στο σημείο αυτό της συζήτησης, το οποίο το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Πρώτος ευχαριστούμε. Αν δεν ζητάει κανένας άλλος το λόγο, ας περάσουμε στην έκθεση... Α, μια κυρία. Η κυρία στο 158. Παρουσιαστείτε παρακαλώ. Γιάνκοβα από την Βουλγαρία, από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Ρατσισμού. Θα ήθελα να ξέρω τι συνέχεια θα δοθεί στις συστάσεις που κάναμε. γιατί το, το εργαστήριο ήταν επιτυχές και πολλοί συνάδελφοι έκαναν πολύ ωραίες προτάσεις. Θα ήθελα να ξέρω πώς θα γυρίσει αυτό με feedback σε εμά αργότερα. Ξέρω ότι μερικές από τις συστάσεις χρειάζονται χρόνο για να υλοποιηθούν. Ερωτώ, είναι δυνατόν να μας πληροφορείτε στο μέλλον για το πώς θα εξελίσσονται τα θέματα αυτά. Πρόεδρος, Κυρία μου, σας προτείνω στο δεύτερο τμήμα να απαντήσουμε συνολικά στο πώς θα δοθεί συνέχεια, όχι μόνο για το δικό σας εργαστήριο, αλλά και για το πρώτο και για το τρίτο. Έτσι ώστε όλοι μαζί από κοινού να δούμε πώς είναι δεπτό να εξασφαλιστεί ένα, ε, μια ενημέρωση σε πάγια βάση, ως συνέχεια να μην μείνει όλο αυτό που συζητήσαμε εδώ ένα ακόμα κείμενο στα χαρτιά όπως τόσο άλλα. Τώρα το λόγο στον εισηγητή του τρίτου εργαστηρίου που έχει το θέμα την πρόσβαση των ατόμων επισφαλούς κατάστασης σε μια πιο διαρκή κατάσταση τρόπου ζωής. Το προέδρευε η κυρία Πακ, δύο συνεισηγητές, η κυρία Μαρή Κριστίν Βερζιά, βουλευτής, και ο κύριος Λουρντέλ της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Σωματείων. Η κυρία Βερζιά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ακούγοντα του συζητητέ των άλλων εργαστηρίων, βλέπω ότι θα έχουμε επικαλύψει σε αυτά που λέμε. Εμεί εστιαστήκαμε κυρίω στην επίπτωση τη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στη ζωή των ατόμων που βρίσκονται σε επισφαλή θέση. Η φτώχεια προϋπήρχε της κρίσης και επιδίνωσε την κατάσταση αυτών που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβασή τους σε ορισμένα δικαιώματα που έχουν. Οι διαφορές μεταξύ των κρατών και στο εσωτερικό των κάθε κράτους υπογραμμίστηκαν στο εργαστήριο. Ορισμένες χώρες, αν δούμε τα νούμερα, φαίνεται ότι τα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι άλλες, γιατί έχουν μεγάλες αποκλήσεις μεταξύ των χωρών. Στατιστικά εννοώ. Μετά είδαμε την ε, ανάγκη λύσεων που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες αυτών των ατόμων που είναι πιο, ιδιαίτερα των πιο τροτών μέσα στην ομάδα αυτή. Σημεία που συζητήθηκαν, το είπαν και τα άλλα εργαστήρια, ήταν το θέμα του εγκάρσιου χαρακτήρα και της ε, ε, ολιστικής, όπως τη λέμε, διάστασης της φτώχειας φαίνεται να μην υπάρχει μια συνολική καθολική πολιτική έναντι των πιο φτωχών στην κοινωνία. Ένα βασικό σημείο είναι το ότι η φτώχεια δεν πρέπει να θεωρείται ως κάτι το μοιραίο και αυτό είναι πρόκληση να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τους πιο φτωχούς. Στο εργαστήριό μας μιλήσαμε για την ανάγκη ευκαμψίας, ευέλικτης δράσης και σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή και είχαμε μαρτυρίες στο εργαστήριο ότι ορισμένοι άνθρωποι που ζουν τραγικές καταστάσεις καταφέρουν να τα φέρουν πέρας, σε πέρας, να τα φέρουν βόλτα. Το ότι είναι φτωχοί και σε τρωτή θέση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουν πλήρη συμμετοχή με τέτοια συζήτηση. Είναι πολίτε με πλήρη δικαιώματα. Όσον αφορά την συλλογική ευκαμψία και ευελιξία, είναι η ματιά που έχουμε έναντι των πιο φτωχών. Πρέπει να τους θεωρούμε ως πλήρει πολίτε, Ιδιαίτερα μου έκανε εντύπωση η μαρτυρία νέων που είχαν διάφορες συναντήσεις και μετέφεραν αυτή τη μαρτυρία Η μαρτυρία έλεγε ότι άτομα λένε αισθανόμαστε να μην υπάρχουμε, κανένα δεν ενδιαφέρεται για μα, γιατί να ενδιαφερθούμε εμεί για άλλου. Άλλο σημείο. Συχνά η φτώχεια θεωρείται μόνο πρόβλημα απασχόλησης. Δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο απασχόλησης και μόνο. Μπορεί κάποιο να βρει δουλειά, παρόλα αυτά να παραμείνει μέσα στην τρωτή ομάδα αν και θα πρέπει να είναι στη θέση να βρει μια απασχόληση. Ένα άτομο δεν είναι μόνο οι σχέσει του με την εργασία. Έχει σημασία η εργασία. Και στο σημείο αυτό υπήρξαν και διαφορετικές απόψεις στο εργαστήριο. Αλλά η κοινωνική αναγνώριση ενός ατόμου χαρακτηρίζεται από πολλές παραμέτρους. Πολλοί τόνισαν την πολιτιστική φερρυπίν διάσταση. Μετά είχαμε το θέμα την πρόσβαση στην εκπαίδευση από όσο πιο μικρή ηλικία γίνεται. Στην Επιτροπή Πολιτισμού ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι στα πρώτα χρόνια της ζωής αποφασίζονται ορισμένα πράγματα για την υπόλοιπη ζωή του ατόμου. Πρόσβαση στην εκπαίδευση λοιπόν, ήδη τα, τα παιδιά από μικρή ηλικία, αλλά και ισόβια κατάρτιση. Οι ανισότητες σε θέματα υγείας και ψυχικής υγείας ιδιαίτερα τονίστηκε και την ανάγκη για μέτρα επίγοντος χαρακτήρα και ειδικών πολιτικών. Όπως και στο εργαστήρι παριθμών 1 και εμείς συζητήσαμε την κατάσταση τροτότητας ορισμένων ομάδων. Αναφέρθηκαν οι γυναίκες που είναι η πλειοψηφία στον πληθυσμό των φτωχών, ιδιαίτερα αυτές που μεγαλώνουν μόνο παιδιά, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, οι ξένοι μετανάστες, παιδιά μεταναστών, ιδιαίτερα αυτοί που προέρχονται από τη Βόρεια Αφρική, από την Μαύρη Αφρική, συγγνώμη. Τέλος, το ότι δεν υπάρχουν κονδύλια επαρκή στον προϋπολογισμό πράγμα το οποίο αποβαίνει σε βάρος των πιο ευπαθών ομάδων, τη στιγμή που σε αυτές τις πολιτικές του κράτους θα έπρεπε ιδιαίτερα να υπάρχει πρόνοια και βοήθεια για τις ευπαθείς ομάδες πολιτιστικά, εκπαίδευση, ε, στο θέμα του σχολείου, η υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, διάφορες ενισχύσεις στις ενώσεις που βοηθάνε αυτές τις ομάδες του πληθυσμού. Αυτά είχα να πω και συνοψίζοντας, εγώ αυτό που ένιωσα μέσα στο εργαστήριο αυτό, την πρόκληση είναι να φροντίσουμε να δοθεί ζωή στην χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, διότι οι ευπαθείς είναι αυτοί που στερούνται ακριβώς αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα και να θεωρούνται τα άτομα αυτά πλήρεις πολίτες. Το είπαν και άλλοι στις παρεμβάσεις τους. Επειδή τα πονάω τα ανθρώπινα δικαιώματα, γι' αυτό τελειώνω με αυτή τη φράση και δίνω το λόγο στον συνεισηγητή μου. Συνεισηγητή μας, ίσως έχει και αυτός να προσθέσει επικοδομητικά σχόλια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στη δικιά μου ομάδα εργασίας, που όπως είπε και η Μαρή Κριστίνα είχαμε μια πλούσια ανταλλαγή απόψεων, καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα, κάποιες προτάσεις που σας μεταφέρουμε εδώ σήμερα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε πολιτικές λαμβάνοντας υπόψη τους πιο φτωχούς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υιοθετούνται μέτρα πολύ συγκεκριμένα για αυτούς, υπέρ αυτών. Σημαίνει επίσης ότι πρέπει να έχουμε οδηγίες, έναν οδικό χάρτη, με συγκεκριμένους στόχους και με συγκεκριμένους επίσης δείκτες που να δείχνουν κατά πόσο καταπολεμάμε όντως τη φτώχεια με τα μέτρα που παίρνουμε και η αξιολόγηση να γίνεται κάθε χρόνο. Επιμείναμε επίσης στο ότι πρέπει να υπάρχει και μια οριζόντια κοινωνική ρήτρα σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε πραγματικό διάλογο με εκείνους που έχουν χαμηλότερα έσοδα, με τους κοινωνικούς εταίρους και με τους διάφορους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Θέλουμε οι εργασίες και τα συμπεράσματα της αγοράς αυτής να ληφθούν υπόψη για την προετοιμασία της επόμενης Ευρωπαϊκής Συνάντησης για τα άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και που οργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα άλλο πόρισμα στο οποίο καταλήξαμε ήταν ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ένδια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό διασφαλίζοντας ε, την πρόσβαση των φτωχών στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό, γι' αυτό βασιζόμαστε και στην έκθεση που υπάρχει για αυτό το θέμα. Κάτι άλλο είναι ότι πρέπει να βγούμε από τη λογική του ανταγωνισμού μεταξύ των ανθρώπων που πλήττονται από τη φτώχεια. Και αυτό θα γίνει κυρίως ε, αλλάζοντας τους μηχανισμούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μηχανισμοί οι οποίοι βασίζονται σε λογικές αμοιβόμενης εργασίας και που τελικά υποφολούνται περισσότερο αυτοί που βρίσκονται μακριά από την αγορά εργασίας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης τον ρόλο των οργανώσεων που δουλεύουν σε αυτό το τομέα, να τις στηρίξουμε οικονομικά και να ε, δώσουμε σημασία στις βέλτιστες πρακτικές. Το ίδιο και για όλους τους φορείς που δρούν στον τομέα αυτό, είτε με μικροπιστώσεις, και να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση και να τους δώσουμε το ευρωπαϊκό καθεστώς. Πρέπει επίσης να φροντίσουμε να υπάρχουν θέσεις απασχόλησης ποιότητας, δηλαδή όχι επισφαλής εργασία. Εδώ βέβαια θέλουμε για τη βοήθεια των κοινωνικών εταίρων αλλά και των κυβερνήσεων. Επίσης το θέμα του φύλου, να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ των δύο φύλων και έγινε μία πρόταση συγκεκριμένη. Οι διαφορές στους μισθούς που υπάρχουν μεταξύ αντρών και γυναικών να μειώνονται κάθε χρόνο 1%. και να δούμε και τα κοινωνικά δικαιώματα για κάθε άτομο. Κάτι άλλο που ζήτησε η ομάδα μας είναι βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών θεσμικών οργάνων υπέρ της καταπολέμησης της φτώχειας. Γιατί η καταπολέμηση της φτώχειας δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα ενός επιτρόπου. Επίσης θέλουμε να υπάρχει καλύτερο συντονισμός μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών, των κοινωνικών υπηρεσιών με εκείνων που ασχολούνται με την υγεία και την εκπαίδευση. Και τέλος, αλλά και λιγότερο σημαντικό, να βάλουμε τον πολίτη σε όποια κοινωνική κατάσταση και αν βρίσκεται, να βάλουμε τον πολίτη λοιπόν στο κέντρο των πολιτικών και των ανησυχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Λουρντέλ. μεγαλώνει η λίστα των συστάσεων και σωστό βεβαίω, αυτό ήταν ο στόχο των εργασιών μα. επειδή πρόκειται για το ίδιο θέμα, α, μήπως θέλετε να λάβετε το λόγο πρώτα εσείς, αλλιώς θα έδινα το λόγο στην διάσκεψη τη συνένεσης που έχει το ίδιο αντικείμενο με το ΤΕΔΙΕ 3, με το εργαστήρι 3. Και μετά να μπορέσουμε να αντιδράσουμε σε όλα αυτά, να παρέμβουμε δηλαδή για όλα αυτά τα θέματα μαζί. ο Ζερόμ Γκίνιον, που προείδρευσε για δυόμιση μέρες την, στην, της διάσκεψης ε, της συνένεσης με κάποιος διακόπτη χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούμε τι λέει. Μέχρι τώρα στις δύο προηγούμενες ομάδες, δηλαδή στους συμμετέχοντές τους, επιτρέψατε να σχολιάσουν την αναφορά των εισηγητών. Θεωρώ ότι είναι δίκαιο και τα μέλη της ομάδας 3 να μπορέσουν να σχολιάσουν τη σχετική αναφορά πριν να προχωρήσετε στην διάσκεψη της συνέντευξης. Μην ανησυχείτε, έχουμε χρόνο. Καλώς λοιπόν. Δίνω το λόγο πρώτα στα μέλη της, του εργαστηρίου 3. Ποιος θέλει το λόγο. Η ΣΕΖ, Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Καλά λοιπόν η κυρία πρώτη. Εγώ είμαι μέλος της Ευρωπαϊκής, και, και, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και θέλω να τονίσω ένα θέμα που συζητήθηκε χθε και που νομίζω ότι δεν περιλαμβάνεται αρκετά ξεκάθαρα στις συστάσεις που ακούσαμε. Δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη δομών που να φέρουν την κοινωνία των πολιτών σε άμεση διασύνδεση με την Ευρωβουλή. Ο στόχος είναι, βέβαια, να εμφανιστούν διάφορες πτυχές της φτώχειας, οι διάφορες καταστάσεις προκαλεί. Αλλά αυτό θα πρέπει να είναι όμως κάτι το τακτικό, όχι επειδή βρισκόμαστε σε κρίση. Η νέα συνθήκη μας δίνει το δικαίωμα αυτό και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να το ακούσει, να το προσέξει αυτό. Να κάνει λοιπόν τακτικές διαβουλεύσεις και στο τέλος να γίνεται μια αγορά των πολιτών όπως αυτή εδώ που να είναι η ολοκλήρωση αυτών των ε, συζητήσεων, αυτών των προσπάθειων. Δεν αρκεί να μιλούμε μονάχα για εθνικές διαδικασίες διαβουλεύσεων. Συχνά στο εθνικό επίπεδο, στο επίπεδο του κράτους μέλους, αγνοούν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Χρειάζεται λοιπόν μια διασύνδεση με τις ε, εργασίες της Ευρωβουλής και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, την οποία εκπροσωπώ. Χρειαζόμαστε πιο ε, σαφείς λοιπόν ε, διασυνδέσεις. Και επίσης υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να διαγραφεί σε ένα από τα σημεία εκεί στις παραγράφους της πρώτης δηλαδή λέει για Black Africa, για Μαύρη Αφρική. Αυτό δεν είναι σωστός όρος και πρέπει να διαγραφεί. Ο κ. Βαν Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τονίζω ένα θέμα στην κατά τα άλλα θαυμάσια ε, σύνοψη που έκανε η, η συγγήτρια. Ενώ το σχολείο. Είμαστε το μόνο εργαστήρι που έδωσε τόση έμφαση στη σχολική εκπαίδευση. Που και προληπτικό χαρακτήρα έχει αλλά και διαρκεί. Θα ήταν σωστό η αγορά να συμμετάσχει στον αγώνα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για να αυξηθούν οι αρμοδιότητες του ευρωπαϊκού επίπεδου για τη βελτίωση της σχολικής εκπαίδευσης. Όπως ξέρετε, τα σχολεία και η εκπαίδευση δεν περιλαμβάνονται μέσα στη συνθήκη. Θεωρούνται ότι είναι καθαρά εθνικά θέματα. Αλλά η Ευρώπη του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα να αναλάβουμε και δράσεις παρακολούθησης αυτού του πάρα πολύ σημαντικού τομέα της ζωής. Όπως η κυρία Βερζιά είπε πριν, υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις χώρες μέλη και υπάρχουν οι πιο καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολύ για να βελτιώσουν την κατάσταση και σε άλλες χώρες που βρίσκονται σε κάποια ε, υστέρηση. Εάν λοιπόν μπορείτε να συμβάλλετε στην προσπάθειά μας να βάλουμε τη σχολική, εκπαίδευση σε ψηλή προτεραιότητα στις λίστες των πραγμάτων που θέλει να κάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εσείς κυρία μου, στο 192. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρο βεβαίω του δύο εινησυγητέ για τη θαυμάσια εργασία που έκαναν. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να τονίσω ένα θέμα με ιδιαίτερη έμφαση που το τόνισα και χθε αλλά νομίζω δεν καλύφθηκε απολύτω στις συστάσεις που μας διάβασαν. Εγώ εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών και τη Συνομοσπονδία Ενώσεων Γυναικών. Έχουμε εδώ μια παράγραφο, τέταρτη πριν από το τέλος, που λέει για την διάσταση της ισότητας του φύλου και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για βελτίωση, ε, για παράδειγμα, Πρέπει να μειωθεί δηλαδή το χάσμα ανάμεσα στις αμοιβές ανθρώπων και γυναικών. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον οι γυναίκες έχουν πρόσβαση σε ποιοτικέ δουλειές, σε δουλειές ποιότητας. Αυτό λέω λοιπόν να, να γράψουμε. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει τις χώρες μέλη για να λάβουν μέτρα σε συνολική διάσταση του προβλήματος ώστε οι γυναίκες που είναι και η πλειοψηφούσα ομάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν τη δυνατότητα να καταλαμβάνουν καλύτερες ε, θέσεις εργασίας. Ακόμα και όταν υπάρχει ε, επαρκής απασχόληση, οι γυναίκες αμείβονται χειρότερα, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν οι σχετικές δομές. Τα ε, σχολεία, για παράδειγμα, τελειώνουν τα μαθήματα στη μία το μεσημέρι. Και επειδή δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί και τέτοια, πρέπει οι γυναίκε να διακόψουν την εργασία του. Άρα δεν μπορούν να δουλεύουν μόνο μέχρι εκείνη την ώρα. Χρειάζονται επομένω δομέ υποστήριξη των γυναικών. Γιατί ε, έτσι όπω είναι με τι ελλείψει αυτέ τώρα, οι γυναίκε βρίσκονται πάντοτε πιο κοντά στα όρια τη φτώχεια. Είναι σημαντική η ανησυχία αυτή και βεβαίω, όπω σα είπα, ανησυχεί ιδίω τι γυναίκε που είναι και οι περισσότερε μέσα στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Το 146. Ο κύριος που είναι στο 146. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ορισμένα πράγματα παραλήφθηκαν από την αναφορά που μας έκανε οι δύο συνεισηγητές. Θέματα τα οποία τονίστηκαν ιδιαίτερα στις συζητήσεις μας χθες. Το πρώτο βέβαια το είπε στην προφορική της σύνοψη η συγγήτρια, αλλά δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο. Δηλαδή ότι πολλοί είπαν ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο απειλείται και ότι αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. Το είπε η συγγήτρια προφορικά, αλλά δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο που τελικά ε, εγκρίναμε. Και μαζί με αυτό και ορισμένες παρεμβάσεις έντονου χαρακτήρα εχθές, ότι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δοθεί πολύ βάρος στην οικονομική διάσταση και όχι αρκετό βάρος στην κοινωνική διάσταση. Και χρειάζεται να υπάρχει κάποια ισορροπία, διότι στην πραγματικότητα αυτά είναι οι δύο πλευρές της ίδιας κατάστασης. Χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη, αλλά χρειάζεται και κοινωνική ανάπτυξη. Και η μία χρειάζεται την άλλη. Ένα άλλο θέμα που δεν φαίνεται τόσο καθαρά στην έκθεση είναι ότι εκφράστηκε πολύ θυμός, πολύ αγανάκτηση στο εργαστήρι σχετικά με την άρνηση των θεσμικών οργάνων της Ευρώπης να αναγνωρίσουν ότι ορισμένες από τις, ορισμένα μέρος από την ευθύνη μάλλον για την κρίση που πλήττει τώρα την Ευρώπη με διάφορους τρόπους ότι ορισμένες λοιπόν από τις ευθύνες αυτές βαρύνουν το ίδιο το ευρωπαϊκό επίπεδο. Όχι βέβαια δεν προκλήθηκαν οι κρίσεις αυτές μόνο από ανόητους χειρισμούς ανόητων ανθρώπων σε ορισμένες περιφερειακές χώρες, αλλά και από λάθο χειρισμού στο επίπεδο της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που προσπάθησαν ε, να προστατεύσουν τις τράπεζες και τους μεγάλους μετόχους τους οι οποίοι έπαιξαν τα χρήματά τους και έχασαν και ξέχασαν την προστασία των πολιτών. Αυτά τα είπαν πολλοί χθε από αυτούς που συμμετείχαν στο εργαστήρι και εγώ θα ήθελα να μπει στο κείμενο. Ένα επίσης πρόσθετο ε, θέμα για το ζήτημα δηλαδή του ελάχιστου εισοδήματος που επίσης ε, συζητήθηκε και στο εργαστήρι παριθμών 1 έγινε μια συγκεκριμένη πρόταση που πάλι δεν περιλήφθηκε εδώ και ήταν η εξή. Η Ευρωβουλή ενδεχομένως και η Κοινωνική και, Οικονομική και η Κοινωνική Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να, να φτιάξουν ένα σύστημα εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματο σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι 50 τώρα χρόνια και παραπάνω μετά από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τότε το 1957 ακόμα υπάρχουν τεράστια ελλείμματα στο θέμα αυτό. Και ένα τελευταίο πράγμα θα ήταν χρήσιμο να συνταχθεί ένας χάρτης που να δομήσει ένα διάλογο ανάμεσα στις οργανώσεις της, κοινωνικής, της κοινωνίας των πολιτών και των οργανισμών της Ευρώπης, των οργάνων της Ευρώπης. Αυτό βεβαίω α το εξετάσει όποιο είναι αρμόδιος. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ για τις ε, παρατηρήσεις σα, Ο κύριος του 234. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, εισηγητές για το ότι συμπεράλαβαν την πρότασή μου στις συστάσεις. Θα είμαι σύντομο γιατί ο προηγούμενο ομιλητή αναφέρθηκε σε αυτό που σκόπευα να πω για τι τράπεζε. Μία σύσταση μόνο. Κάτι που δεν είπα χθε στο εργαστήριο. Εγώ είμαι Βούλγαρος. Η χώρα είναι υπό το μηχανισμό επαπτείας, λεγόμενος μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου η σύστασή μου και θα σας φέρνει λίγο περίεργο γιατί δεν ισχύει για τις περισσότερες άλλες χώρες ό,τι μέτρα και να πάρουμε εθνικά ή ευρωπαϊκά δεν θα είναι αποδοτικά αν δεν είναι διαφανή και αν δεν χαρακτηρίζονται από υπολογία. Γιατί η διαφθορά, η οικονομική διαφθορά εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μου και θα ήθελα να αναφερθεί ρητά ότι ό,τι μέτρα οι πολιτικές εφαρμοστούν είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο η αρχή της διαφάνειας και της ευθύνης θα πρέπει να εφαρμόζεται. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το σχόλιο. Ακόμα και ό,τι ακούμε μετά το εργαστήριο θα τα βάλουμε σε παράρτημα. η διέκθεση έχει εγκριθεί, δεν μπορούν να μπουν αλλά δεν θα πάνε χαμένες, ε, θα μπουν σε παράρτημα. 281. Η κυρία Ρελιού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους δύο συγγητέ και μία διευκρινήση για το σημείο 5. Η αναγνώριση της σχέσης με τις άκρας φτώχειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ευρωκοινοβούλιο το 2008 ψήφισε την έκθεση Κάσμαν προκειμένου να μπει ο όρος του κοινωνικού αποκλεισμού και της άκρας πτώχειας στο πολιετές πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ας πάρουμε την απόφαση αυτή του Ευρωκοινοβουλίου που δυστυχώς την απέρριψε το Συμβούλιο. Ας πάρουμε αυτό που ήδη υπάρχει για να υποστηριχθεί το αίτημα για μια μελέτη στα πλαίσια πολιετούς μελέτης στο μέλλον. Και η μελέτη αυτή να γίνει σε συνεργασία με τα άτομα που ζουν αυτή την κατάσταση, να μην είναι μόνο μια μελέτη εμπειρογνωμόνων, αλλά με άτομα που ζουν αυτή την κατάσταση και που θα δώσουν στους άλλους να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται και πώς είναι δυνατόν να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. ο αριθμός 331, ο κύριος. Από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέχνων Ελλάδος. Μια πρώτη παρατήρηση, επειδή η οικονομική κρίση πλήττει εκτός από τα άτομα και τις οικογένειες, θέλω να παρακαλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει την πρωτοβουλία για αλλαγή του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, έτσι ώστε να γίνει υποχρεωτική για κάθε κράτος μέλος η τοποθέτηση ενός εκ των μελών κάθε κράτους μέλους για να προέρχεται από τη μεγαλύτερη οικογενειακή οργάνωση κάθε κράτους μέλους. Θέλουμε δηλαδή στην ομάδα 3 υποχρεωτικά να υπάρχει ένας εκπρόσωπος από οικογενειακή οργάνωση από κάθε κράτος μέλος, έτσι ώστε η φωνή της οικογένειας να ακούγεται μέσω της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Ένα δεύτερο σχόλιο που αφορά και τα τρία εργαστήρια έχει σχέση με τις πολίτεκνες, τις μεγάλες οικογένειες. Οι οικογένειες που έχουν πολλά παιδιά πλήττονται αναλογικά περισσότερο λόγω της κρίσης από τους άμεσους και έμεσους φόρους. Και βέβαια υπάρχουν κείμενα στην Ευρώπη που αναγνωρίζουν τις πολίτεχνες οικογένειες ως ευπαθής κοινωνική ομάδα. Ειδικότερα όμως στις χώρες που έχουν μέτρα λιτότητας παρατηρούμε ότι περικόπτονται ή μειώνονται σημαντικά τα επιδόματα των παιδιών, ενώ από την άλλη μεριά αυξάνονται αναγκαστικά τα χρηματικά κονδύλια που αφορούν νόμιμους ή μη νόμιμους μετανάστες. Αυτό δυστυχώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις δημιουργίας ξενοφοβίας και ρατσισμού σε μερικά κράτη. Το σημείο αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να είχε τύχει περισσότερης προσοχής και ανάλυσης στα εργαστήρια και θα έπρεπε να υπάρξει μια τοποθέτηση και από εσά το Προεδρείο αλλά και γενικότερα της αγοράς σχετικά με την περικοπή των επιδομάτων των παιδιών και γενικότερα των κονδυλίων που αφορούν τη στήριξη της οικογένειας τώρα που βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης ή ακόμα περισσότερο στα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν προγράμματα λιτότητας. Ευχαριστώ. Ε, Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε. ο κύριος Μελισσιάς της ΟΚΕ. Θα επανέλθουμε μετά, έχω ακόμα μία παρέμβαση, μετά θα, θα επανέλθουμε στο τέλος της συζήτησης. Μελίσιας λέγομαι. Χαίρομαι για την υλοποίηση αυτή τη αγορά, τη διεξαγωγή αυτή τη συνεδρίαση δηλαδή, που αποτελεί συμμετοχή, επιτρέπει τη συμμετοχή, δηλαδή την άμεση συμμετοχή των οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών. Τονίζω εδώ ότι είναι σημαντικό το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί παραπέρα. Στην τρίτη παύλα, αυτό λέω, και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση υπερασπιζόμενοι και τις βασικές αρχές μας, δηλαδή το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ιδέα της συλλογική ευθύνης και της αλληλεγγύης. Η φτώχεια είναι το πρόβλημα, αλλά όχι μόνο των φτωχών. Γι' αυτό τονίζω και πάλι ότι έχει ο καθένας το δικαίωμα να μην αφαιθεί μοναχός του στην τύχη του μέσα στην κρίση. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει σημαντικές αρμοδιότητες. Στην διάρκεια της τελευταίας ολομέλειας συζητήθηκε η φτώχεια και τα τρόφιμα, η έλλειψη τροφίμων. Υπάρχουν όμως και άλλα. Υπάρχει η φτώχεια που δεν επιτρέπει σε κάποιον να, έχει, να μπορεί να ε, έχει στη διάθεσή του επαρκή ενέργεια, ηλεκτρικό ρεύμα για παράδειγμα, πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Ε, σε αυτά προστίθεται και η δημογραφική κρίση. Τα βλέπουμε αυτά, για παράδειγμα, στην Ισπανία. Πρέπει να αποφευχθεί τελικά και η φτώχεια της αλληλεγγύης, δηλαδή να υπάρξει έλλειμμα αλληλεγγύης. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν συνεργασίες, να γίνουν συμφωνίες, τα είπαμε αυτά εχθές ο δημόσιος τομέας να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Τέτοιες συνεργασίες υπάρχουν για παράδειγμα στη χώρα μου την Πορτογαλία. Επίσης σημαντικό είναι να αποφευθεί η υπερχρέωση των οικογενειών. Βλέπουμε για παράδειγμα στην κεντρική Ιταλία, στην Τοσκάνη, όπου κράτος, εκκλησία, τράπεζες κοινωνικές οργανώσεις όπως η Μισερικόρδια συνεργάζονται για να προσφέρουν βοήθεια σε αυτούς που θίγονται περισσότερο. Οι οργανώσεις που εκπροσωπούνται και σήμερα εδώ πρέπει να ασκήσουν πίεση στην κατεύθυνση αυτή. Και θα έρθω και σε κάτι που ακούστηκε από άλλο εργαστήριο, δηλαδή το εξασφαλισμένο, το εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα. Στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή πριν από δύο χρόνια είχαμε μία έκθεση για το άσυλο και είχε θέσει και το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. 342 εσείς κυρία μου. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ για τη σύσταση που λέει ότι πρέπει να περιλαμβάνονται και οι γνώμες, να ακούγονται μάλλον οι άνθρωποι που θίγονται περισσότερο από τη φτώχεια. Αυτό δεν είναι απλώς θέμα ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να έχετε καλές προτάσεις λύσεων εάν δεν ακούσετε τους άμεσα θυγόμενους. Στο 4 τώρα δεν οργανώνονται, έχει υπάρχει μια, ένα σφάλμα, δεν οργανώνονται από το κοινοβούλιο οι αιτήσει συναντήσεις των ε, ε, οργανώσεων αυτών με τα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά από την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Και τα, οργανώνουμε, τα οργανώνουμε εδώ και 10 χρόνια από το 2001. Και με οργανώσεις οι οποίες ε, συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή και η παρακολούθηση γίνεται μετά μετά σε ολόκληρο το χρόνο. Θα έπρεπε λοιπόν να πούμε εδώ να διασφαλιστεί μία διασύνδεση μεταξύ εθνικών και ε, ευρωπαϊκών οργανώσεων και για τα πρόσωπα, δηλαδή για την προσώπηση των προσώπων που θίγονται πολύ από τη φτώχεια. Ευχαριστώ για την διευκρίνηση αυτή, για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και συνδιασκέψεις. Το 229. Δεν γνωρίζω τα ονόματα. Κάποια μιλάει χωρίς μικρόφωνο. Madame, je vous invite à donner votre nom, mais moi je ne le connais pas, donc je ne peux pas vous appeler par votre nom puisque je ne le connais pas. Mais je vous demande alors de vous présenter. Δεν γνωρίζω το όνομά σας, δεν μπορώ λοιπόν να σας αποκαλέσω με το όνομά σας. Παρακαλώ λοιπόν αυτό συστηθείτε, απαντάει η Πρόεδρος. Ορίστε παρακαλώ. Εσείς, εσείς. Νομίζω, νομίζω ότι είχατε πει 229. Πραγματικά ε, θεωρώ τις δύο αυτές μέρες εξαιρετικά σημαντικές, όπως είπα και χτες, και νομίζω ότι ήταν σημαντικό το ότι αυτή η θεσμική, θα έλεγα, παρέμβαση ε, έχει τη μεγάλη της αξία. Ποια είναι όμως η ποιοτική διαφορά πάνω σε αυτό. Χτες και στο εργαστήριο 3, το οποίο απεικονίζεται αλλά όχι με πάρα πολύ έντονο τρόπο, μιλήσαμε πάρα πολύ για το το, ότι η ευρώπη σήμερα σύμφωνα με τις απόψεις των πολιτών της και φαντάζομαι ότι αυτό το εκπροσωπεί περισσότερο από, από κάθε άλλο όργανο ε, το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο μιλήσαμε λοιπόν ότι εκείνο που κινδυνεύει αυτή τη στιγμή είναι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο το οποίο βεβαίως συνθλίβει εάν εξακολουθήσει να μην ε, αλλάξει η πορεία συνθλίβει τους πολίτες. εγώ ε, εκπροσωπώ όπως είπα την ελληνική αντιπροσωπεία είμαι ε, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας του ευρωπαϊκού λόμπι γυναικών σε μια χώρα που σήμερα πραγματικά πλήττεται βαριά και έχει μπει σε μια ε, κατάσταση και τόσο μέσω του διεθνούς νομισματικού ταμείου όσο και της εποπτείας της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία ενδεχομένως έχει πολλά σημαντικά στοιχεία αλλά εκείνο που διαλύει πραγματικά είναι ε, η ελληνίδα και ο έλληνας πολίτης. εκατοντάδες άνεργοι προστίθενται καθημερινά σε αυτούς που ήδη υπάρχουν. θεωρώ ότι πλέον το μοντέλο αυτό δεν θα μπορέσει να ωφελήσει τη χώρα αν δεν προσαρμοστεί στις αρχές και τις αξίες οι οποίες είναι η αλληλεγγύη η ίση μεταχείριση αλλά κυρίως το γεγονός ότι σήμερα την κρίση την πληρώνουν και στη χώρα μου οι πλέον ευάλωτες ομάδες. μιλάμε πολύ σωστά ότι η φτώχεια αποτελεί έλλειψη κοινωνικού ε, ερίσματος. δεν έχουμε σήμερα το δικαίωμα να αφήσουμε απροστάτευτους τους πολίτες κάθε χώρας η οποία υφίσταται ενδεχομένως ε, ε, τα αποτελέσματα μιας κρίσης στην οποία ελάχιστα συνέβαλε. Και αν αυτό το κοινωνικό μοντέλο δεν καταφέρουμε να το σώσουμε με θεσμούς, με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, με αλληλεγγύη και αλληλοσεβασμό, τότε η Ευρώπη δεν, δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό είναι το κυρίως ε, το κύριο θέμα σήμερα και αυτή είναι η ποιοτική παρέμβαση που πραγματικά πιστεύω ότι το, ε, αυτή η, η συνάντηση πρέπει να φέρει επίσης σαν μήνυμα και ενώνω φωνές ε, μου, τη φωνή μου με εκείνους που είπαν πραγματικά ότι αυτό που αξίζει να διασώσουμε είναι η Ευρώπη και η Ευρώπη εδώ και 50 χρόνια στήθηκε πάνω στον άνθρωπο με κέντρο τον άνθρωπο. Είναι, μεγάλο, είναι μεγάλη η ευθύνη που αυτή τη στιγμή βαρύνει όλους μας, αλλά εμείς οι πολίτες θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Και σε εσά εναποθέτουμε τις ελπίδες μας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το συνολικό ολοκληρωμένο μήνυμα. Ακόμη ζητούν ορισμένοι να τους επιτρέπει μια παρέμβαση σε ορισμένους αριθμούς θέσεων, δεν γνωρίζω τα ονόματα. Θα σας δώσω τον λόγο μετά, θα δώσω τον λόγο τώρα στους πολίτες και αμέσως μετά το διάλειμμα θα σας δώσω τον λόγο στα πρόσωπα που ε, ανέφερα προηγουμένως και που έχουν ήδη ζητήσει το λόγο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βινιό που συντόνισε το έργο των 20 πολιτών που έχουν έλθει από 15 ε, διαφορετικές χώρες μέλη και που εργάστηκαν για έναν αριθμό θεμάτων. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Ζερόμ Βινιού. Είχα την τύχη να προεδρεύω δύο μέρες την διάσκεψη της συνένεσης που κλήθηκε να φέρει αποτελέσματα, να καταλήξει σε συμφωνία, σε συνένεση πάνω σε προτάσεις που δίνουν απαντήσεις στις δύο ερωτήσεις που τους στέθηκαν. Πρώτη ερώτηση. Τι μέτρα και τι δράσεις πρέπει να ληφθούν προκειμένου οι ηλικιωμένοι και χαμηλών εισοδημάτων να μπορούν να έχουν πιο εύκολα πρόσβαση στον πολιτισμό και στις νέες τεχνολογίες. Δεύτερη ερώτηση ήταν τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλος ιδιαίτερος τι μέτρα και τι δράσεις πρέπει να αναλάβει για να πετύχει αυτό. Τα πορίσματα των εργασιών αυτών, οι προτάσεις, εγκρίθηκαν στην ομάδα μας με συνένεση και θα σας παρουσιαστούν από τη Μαρία Καμπρέν για τον πολιτισμό και από τον Άλμπερ Φιναμπεδεφέλτ για τις νέες τεχνολογίες. Ως πρόεδρος της ομάδας αυτής θέλω να σας μεταφέρω τον δυνατιστώσαμε στην προσπάθειά μας αυτή και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ανέλαβε την πρωτοβουλία. Βλέπετε, ξεκινήσαμε από μία διαμαρτυρία, από δυσαρέσκεια. Γιατί μας είπανε πώς μας λέτε να καθίσουμε να σκεφτούμε την πρόσβαση στον πολιτισμό όταν οι συντάξει σε μερικές χώρες είναι τόσο χαμηλές, πώς είναι δυνατόν να μας λέτε για πρόσβαση στον πολιτισμό όταν πολιτισμός δεν υπάρχει στην καθημερινή μας ζωή. Και σε ορισμένες χώρες ε, είπαν ότι ορισμένοι θα προτιμούσαν οι γέροι να είχαν πεθάνει. Πώς είναι δυνατόν να μας μιλάτε, μου είπανε, για πρόσβαση στον πολιτισμό όταν, ή στι νέε τεχνολογίες, όταν δεν έχουμε καθόλου εξυγχρονισμό και όταν ε, ο κομμουνισμός στον οποίο ζήσαμε και μεγαλώσαμε είναι κάτι που πρέπει να ξεχάσουμε. Αυτή η οργή, αυτή η αγανάκτηση σιγά σιγά διοχετεύτηκε σε προτάσεις. Αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, έτσι είπε κάποιος. Είναι ένας φαύλος κύκλος όταν από τη μια μεριά έχουμε τις ανισότητες που δημιουργούν φτώχεια και η φτώχεια δημιουργεί την αναδίπλωση στον εαυτό μας και η αναδίπλωση στον εαυτό μας σημαίνει έλλειψη αλληλεγγύης και χωρίς αλληλεγγύη δεν έχουμε την πολιτική δύναμη να προχωρήσουμε σε λύσει. Για να βγούμε λοιπόν από αυτό το φαύλο κύκλο πρέπει να γίνει κάτι και από τι δύο πλευρέ. Και από αυτού που λέμε ότι είναι πλούσιοι και από αυτού που λέμε ότι είναι φτωχοί και απομονωμένοι. Υπάρχει δυνατότητα, αν γίνουν προσπάθειες και από τις δύο πλευρές, να πάμε μπροστά. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στη Μαρία Καμπράλ καταρχήν για να μας μιλήσει για τα μέτρα που προτείνουμε όσον αφορά την πρόσβαση στον πολιτισμό. Ευχαριστώ. Πρώτο σημείο. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την ευημερία και το επίπεδο ζωής. Οι συντάξει πρέπει να προσαρμόζονται στο κόστος ζωής και δεν πρέπει να υποβάλλονται σε φορολόγηση. Προκειμένου να βελτιώσουμε την κατανόηση, να μας καταλάβουν καλύτερα δηλαδή οι πολιτικά ηθήνοντες, θα πρέπει οι πολιτικές που έχουν να κάνουν με την ένδια και με τους ηλικιωμένου να φροντίσουμε οι θύνοντες αυτοί οι πολιτικοί να περνάνε ένα μέρος της ζωής τους κάθε χρόνο κοντά στους πιο φτωχούς για να συνειδητοποιήσουν τι επιπτώσεις έχει η πολιτική που αποφασίζουν επί τόπου, πάνω στους φτωχούς. Οι ηλικιωμένοι από την άλλη αποτελούν ένα, μια πηγή, ένα πλούτο γνώσης και πολύτιμη εμπειρίας για το σύνολο της κοινωνίας. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να δώσουν μεγάλη θέση στη δημιουργία και να μην κλείνουν οι δομές οι οποίες διευκολύνουν τις επαφές ανάμεσα στις πιο νέες γενιές και τους ηλικιωμένους όπως να υπάρχουν για παράδειγμα κατοικίες όπου να, να ζουν και νέοι και ηλικιωμένοι, να υπάρχουν κέντρα υποδοχής ηλικιωμένων. Έπειτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη πρέπει να φροντίσουν και για την πλήρη απασχόληση αλλά και για την πλήρη δραστηριότητα. Δηλαδή, προτείνουμε η μεταρρύθμιση των συντονιστών να γίνει ώστε να συνδυάσει τι συντάξεις με άλλες πηγές εισοδημάτων από άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα τον εθελοντισμό. Επίτα, για να πετύχουμε συνθήκες ε, ζωής ικανοποιητικές για τους πιο ευάλωτους ηλικιωμένους, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να υιοθετούν μέτρα μείωσης του κόστους, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αγαθά και οι φτωχοί ηλικιωμένοι και η πρόσβαση στα, να υπάρχει πρόσβαση σε πιστώσεις για την υγεία ή για τη στέγαση που να μην στοιχίζουν πιο ακριβά για τους πιο φτωχούς από ό,τι για τους λιγότερο φτωχούς. Έπειτα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να φροντίσουν να διασφαλίσουν αποτελεσματική πρόσβαση σε όλα τα αγαθά και στα πολιτιστικά αγαθά, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν στη μετακίνηση ηλικιωμένοι. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσφέρει μία πλατφόρμα ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να μαζεύονται και να ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν ώστε με τη σειρά του άλλα κράτη να μπορούν και αυτά να τις εφαρμόσουν. Ευχαριστώ πολύ. Η Αλμπερτίνα τώρα θα παρουσιάσει τις ε, προτάσεις μας όσον αφορά την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Προτάσεις τις οποίες καταλήξαμε με συνένεση. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία αυτή. Συζητήσαμε για το ψηφιακό χάσμα. Προτάσεις μας είναι οι εξής. Όλοι οι άνθρωποι δυσκολεύονται για τη, στη χρήση νέων τεχνολογιών είτε λόγω της γλώσσας που χρησιμοποιείται στα μαθήματα που δεν μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε είτε για άλλους λόγους. Οι ηλικιωμένοι δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Κάτι το οποίο θα ήταν ε, αναγκαίο για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε παρετέρω κατάρτιση. Έπειτα, πρέπει να φροντίσουμε να έχουν πρόσβαση στα μηχανήματα αυτά, στις υποδομές των νέων τεχνολογιών για να μπορέσουν να εξοικειωθούν. Αλλιώς απομονώνονται μην γνωρίζοντας τίποτα για την ψηφιακή τεχνολογία. Γι' αυτό Ευρω... το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να ενθαρρύνει. Να υπάρχουν χώροι, κέντρα, καταστάσεις όπου όλοι οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τίποτα για τις ε, νέες τεχνολογίες και που δεν έχουν πόρους να μπορούν να έχουν ελεύθερα πρόσβαση ώστε να μάθουν για τις νέες τεχνολογίες με μαθήματα τα οποία θα διδάσκουν κατάλληλοι άνθρωποι οι οποίοι θα γνωρίζουν τις δυσκολίες εκμάθησης που έχουν ηλικιωμένοι. Οι εγχειρίδια, τα οποία να πρέπει δηλαδή να φτιάξουμε εγχειρίδια τα οποία να γραφτούν με τρόπο απόλυτα κατανοητό από τους ηλικιωμένους, να είναι προσαρμοσμένα δηλαδή τα εγχειρίδια αυτά στους ηλικιωμένους και στις αδυναμίες ή δυνατότητες που έχουν. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο για το χρήστη τι ακριβώς κάνει σε κάθε βήμα εκμάθησης νέων τεχνολογιών. Συχνά οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Αν οι νέοι λοιπόν θα ήταν καλύτερα ενημερωμένοι, θα μπορούσαν να δείξουν την αλληλεγγύη τους απέναντι στους ηλικιωμένους και να τους μάθουν πολλά πράγματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο σε αυτήν την ε, σχέση, τη σύνδεση ανάμεσα στις διάφορες γενιές ώστε οι νεότερες γενιές να δείξουν την αλληλεγγύη τους προς τους ηλικιωμένου και να μην υπάρχει τέτοιο χάσμα μεταξύ τους. Έπειτα πρέπει οι νέοι να ενημερωθούν. Να ενημερωθούν για το πρόβλημα που έχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι αποκλείονται από την ψηφιακή τεχνολογία. Οι νέοι πρέπει να μπορέσουν να καταλάβουν τις δυσκολίες των ηλικιωμένων και πρέπει να τους ανθαρρύνουμε να είναι θελοντές και να βοηθούν τους ηλικιωμένου. Βλέπετε κάθε νέο μηχάνημα πολύ γρήγορα ε, γίνεται παλιό γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται και προδεύει και είναι δύσκολο οι ηλικιωμένοι να παρακολουθήσουν τις αλλαγές αυτές. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι πολλά ε, μηχανήματα φτιάχνονται ε, με στόχο ως πελάτη το νέο. Οπότε και εκεί δυσκολεύονται οι ηλικιωμένοι. Δεδομένου λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τις νέες γενιές, αλλά πόσο μάλλον για τους ηλικιωμένους να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας πληροφοριών, να είναι ενήμεροι και να αντιλαμβάνονται πώς δουλεύουν τα διάφορα μηχανήματα και δεν έχουν και τους πόρους, θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα να ενθαρρύνει την ανάπτυξη πιο απλών ε, μηχανών και μηχανημάτων τα οποία να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ηλικιωμένων. Βλέπετε, οι φτωχοί, μάλλον για τους φτωχούς, η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες είναι πιο ακριβή από ό,τι για τους υπόλοιπους. Για παράδειγμα, αν αγοράσετε μια κάρτα κινητού, είναι πιο ακριβό το τηλεφώνημα τότε από ότι αν έχεις συνδρομή σε μια τηλεφωνική εταιρεία. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να στηρίξουμε τους ηλικιωμένου ώστε να έχουν πρόσβαση στην κινητή τηλεφωνία στα κομπιούτερ, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές δηλαδή, με φτηνό κόστος. Δεδομένου ότι καμία τεχνολογία δεν μπορεί να βελτιώσει επιτυχώς την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, είναι τελικά ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών να προωθήσουν τις νέες τεχνολογίες και να φροντίσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές οι ηλικιωμένοι, όχι μόνο σαν εργαλείο, αλλά και για να βελτιώσουν το επίπεδο της κοινωνικής του ζωής. Έπειτα έτσι θα έχουν την ευκαιρία να βάλουν και το μυαλό τους να δουλέψει και είναι και μια ευκαιρία να επικοινωνήσουν έτσι περισσότερο με τις οικογένειές τους. Η πρόσβαση στην ε, πληροφορία πρέπει και στην επικοινωνία πρέπει να είναι κάτι πιο φτηνό. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Κύριε Βινιό, ένα μικρό συμπλήρωμα νομίζω. Βινιό, επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο. Όχι πόρισμα, αλλά αναφέρεται στο θέμα της αγοράς. Κρίση και φτώχεια πολύ παρούσα η κρίση και φτώχεια στη συζήτησή μας σε σχέση με την αύξηση του κινδύνου της για φτώχεια όπως επίσης και την, το τι αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν στην ευρωπαϊκή κοινωνία λόγω της κρίσης. Στις συζητήσεις που είχαμε κρίνουμε ότι αναζητούμε κάτι που θα ενώσει τους Ευρωπαίους η κρίση ενδεχομένως προσφέρει τη δυνατότητα να μην ενωθούν μόνο όσον αφορά το τι κατέχουν, τα υπάρχοντά τους, γιατί όταν συχνά όταν αυτή είναι η βάση είναι αμυντική η κίνηση, αλλά να συνενωθούν σε σχέση με το τι τους λείπει. Άρα να υπάρχει μια συμπληρωματικότητα. Οι ηλικιωμένοι, αυτοί που έχουν ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα, έχουν ένα πλούτο μνήμη και χρόνος. Η μνήμη και ο χρόνος λείπουν στους πιο νέους και σε αυτούς που είναι πολύ απορροφημένοι από το επάγγελμα που ασκούν. Άρα, πώς μπορούμε να δούμε ο πλούτος των μεν να καλύψει τις ελλείψεις των άλλων. Αυτό ήταν παρόν στην δουλειά που κάναμε. Ευχαριστώ. Ένας από τους συμμετέχοντες ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ και καλή σας μέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έρχομαι από την Ισπανία εγώ. Δεν εκπροσωπώ καμία οργάνωση, κανένα συνδικάτο, κανένα φόρουμ. Έρχομαι ως άτομο, ως Ισπανός πολίτης εδώ. Πράγματι, σε όλες τις χώρες, από ό,τι βλέπω αυτές τις τρεις μέρες που είμαι εδώ, έχουμε προβλήματα την κρίση, τη φτώχεια, πώς να βγούμε από αυτήν και πώς να έχουμε πρόσβαση στον πολιτισμό και στις νέες τεχνολογίες χωρίς αυτό να μας κοστίζει πολλά λεφτά. Στην συνάντησή μας αυτή, στη συνένεση, δουλέψαμε πάνω σε αυτό το θέμα και δουλέψαμε πάνω σε ένα θέμα το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στα συμπεράσματά μας, που εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Στις χώρες μας, όταν μιλάμε για νέες τεχνολογίες, υπολογιστές, κινητά κτλ. Η γλώσσα των εγχειριδίων είναι τέτοια, μάλλον είναι στα αγγλικά, άντε και στα γαλλικά. Ξέρω ότι υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι σε όλες τις χώρες είναι υποχρεωτικό στις χώρες όπου χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός αυτός ή το προϊόν αυτό να πρέπει να υπάρχει και μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα. Είτε πρόκειται για τα ρουμανικά, είτε τα ελληνικά, είτε τα δεν ξέρω εγώ τι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να φροντίσει να τηρείται πράγματι η νομοθεσία αυτή. Γιατί εμεί που είμαστε πιο μεγάλοι, ηλικιωμένοι, ε, δεν ξέρουμε τόσε πολλέ ξένε γλώσσε όπω ξέρουν οι νέοι σήμερα. Εμεί ηλικιωμένοι δεν έχουμε μάθει ξένε γλώσσε. Έχουμε μάθει τη δικιά μας μόνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ για το συμπληρωματικό σχόλιο. Έτσι προς το παρόν σταματάμε εδώ τις εργασίες μας, θα κάνουμε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά. Και θυμίζω αυτά, αυτούς που ανάφερα και όσοι έστελναν γραπτά ερωτήματα να οργανώσουμε το δεύτερο μέρος της συζήτησης για να κλείσουμε την αγορά αυτή. Μετά το διάλειμμα αυτό για καφέ, σα επισημαίνω ότι μπορείτε τα κείμενα που έχετε για την επιστροφή των οδηπορικών να τα δώσετε στο είσοδο τη αιθούς, θα υπάρχουν δύο άτομα αρμόδια εκεί. όπω επίση βγαίνοντα από το κτίριο μπορείτε να δώσετε έντυπα από την έκθεση Εσπλανάντα από όπου μπήκατε χθε. Γιατί αν δεν δώσετε τα, το, το έντυπο αυτό συμπληρωμένο δεν θα σε επιστραφούν τα χρήματα. Αυτοί που πήραν μέρο στην consensus έχουν πάρει ήδη τι οδηγίες σχετικέ. Τα πιστοποιητικά συμμετοχή θα μοιραστούν στην είσοδο του ημικυκλίου, στο διάλειμμα. Πάρτε τον καφέ σας, θα παρουσιάσουμε τι συστάσει στον τύπο εμεί και σε 15 λεπτά ξαναρχίζουμε. 15-20 λεπτά το πολύ ξαναρχίζουμε.